Να ξεκινήσουμε, συνάδελφοι, και ο Μπράουντο, παρακαλώ να κάτσει. Okay, ich rufe auf den Tagesordnungs... Μάλιστα. Και να πάμε λοιπόν παρά αυτά στο σημείο νέα της ημερήσιας διάταξης ψηφοφορίες. Ξεκινάμε σε ό,τι αφορά έγκριση γνωμοδότηση υπομορφή επιστολή σχετικά με την αίτηση κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού το ταφπί. υπέρ παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε ψηφίζουμε λοιπόν αν ψηφίσατε όλοι πέρας το υπέρ 6 κατά εγκρίνεται. Δεύτερο σούπερ μάρκετ Λαρίσα από την Ελλάδα. Ψηφίζουμε. Gestimmt. Σούπερ μάρκετ Λάρισα. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Επίσης εγκρίθηκε. στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπαιων. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική C, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 τροπολογία υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι μάλλον δεν περνάει, αλλά ας ελέγξουμε παρακαλώ έναρξη ψηφοφορίας. πέρασε. Απορρίπτεται. Η 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 40. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. ψήφισετε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 41 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεργαστική ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά αποχές έγκρινεται 66 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 67 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχο ζητητά έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 68. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Προπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τρία υπέρ μισό λεπτό. Καταπεπτεί η τρία και πάμε στην τέσσερα. Α, πρέπει να ψηφίσουμε και την τρία. Εντάξει λοιπόν. Ζητώ συγγνώμη. Η τρία λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η πέντε, με προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Το individual measures γίνεται individual actors. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η έξι, Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Υπτά. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Άρα το ελέγξουμε. Τη 19. Δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές. Μα τι γίνεται, έχετε κουραστεί, θα σηκώνετε τα χέρια σας. Να ελέγξουμε παρακαλώ τον 28 ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρασε. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 30. Με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Η 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται και τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότηση που πώς τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. 43 υπέρ, 4 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. εφαρμογή τη Σύμβαση του Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με ιδιαίτερη έμφαση στι καταληκτικέ παρατηρήσει τη Επιτροπή του ΟΗΕ. Εξαιρετικό τίτλο. Η Η κυρία Έλικα Στίβεν. Και πρωτού ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει. Σας παρακαλώ ησυχία και οι συζητήσεις έξω. Wir warten einen Moment. Περιμένουμε μισό λεπτό. Ciao, Paloma, please. Ciao, Paloma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 So, dann können wir den Tagesordnung... Μάλιστα, και έτσι λοιπόν στο 12 τη ημερήσιας ε, διάταξη. η συγκεκριμένη κυρία Έλγα Στίβενς και να σα πω ότι θα έχουμε κάποιε εικόνε ε, στην οθόνη θα μοιραστούν οι κάρτε τρει στον καθένα Έχουμε πάλι λοιπόν τις τρεις κάρτες, τις τρεις άγιες κάρτες αυτές. Η πράσινη υποδεικνύει ότι κατανοούμε τον ομιλητή και το μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε. Η κίτρινη κάρτα είναι η κάρτα την οποία μπορούμε να σηκώσουμε αν δεν καταλαβαίνουμε τον ε, ομιλητή ή σε περίπτωση που μιλάει πάρα πολύ γρήγορα και μάλλον αν μιλάει πολύ γρήγορα ο ομιλητής υπάρχει η κόκκινη κάρτα αυτή. Αυτή τη διαδικασία λοιπόν θα ακολουθήσουμε και ελπίζω όλοι να έχετε τις κάρτες σας γιατί αποτελούν τμήμα τη βασικού εξοπλισμού στην Επιτροπή μας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Η Έλκα Στίβενς έχει το λόγο. Πείτε. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις για τη συνεργασία τους. Να ευχαριστήσω επίσης και τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι στην συγκεκριμένη Intergroup έχουν συνυπογράψει πολλές από τις τροπολογίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των τροπολογιών γιατί αν είχαμε να ασχοληθούμε με την κάθε μία ξεχωριστά θα είχαμε πολύ περισσότερη δουλειά. Τώρα έχουμε έναν αριθμό διαχειρίσιμο και να καταλήξουμε ελπίζω εύκολα σε συμβιβαστικές προτάσεις. Να ευχαριστήσω επίσης και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για ΑΜΕΑ για τη συνεργασία του τους τελευταίους μήνες. Να τονίσω εδώ την ευανάγνωστη έκθεση μετά από τη συμπερίληψη των προτάσεών σας. Η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή επίσης μας δίνει την δυνατότητα με τις τρεις κάρτες τις οποίες σας μοιράσαμε να μπορέσετε να κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε. δεν υπάρχει η αυτόματη εφαρμογή από ομιλία σε κείμενο που διευκολύνει κάποιους από μας που έχουμε θέματα, αλλά είναι αλήθεια ότι εκεί που υπάρχει κανένας δεν μπορεί να διαβάσει αυτά τα οποία λέω. Ελπίζω λοιπόν την επόμενη φορά να τα οργανώσουμε καλύτερα έτσι ώστε ε, να ε, γίνεται η ε, η ανάγνωση του, της ομιλίας μου, της ομιλίας του διερμηνέα μου έτσι όπως ακούγεται μετατρέπεται σε κείμενο γραπτό. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αφορά μόνο ε, τα θέματα των αναπηριών. Όλοι οι πολίτες ε, είτε έχουν προβλήματα είτε δεν έχουν πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν συζητήσεις σαν τη δική μας ανεξαρτήτως αν είναι συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής, ολομέλειας, όποιος και αν παρακολουθεί, άνδρες, γυναίκες, ανεξαρτήτως φίλου κτλ. πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις συζητήσεις. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν συνάδελφοι οι συνεδριάσεις μας να είναι εύκολες στην παρακολούθησή τους, δεν είναι δημοσιονομικό το θέμα, το θέμα είναι να το ε, θελήσουμε. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σας ενημερώσω λίγο για τις τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες θα τις στείλει το γραφείο μου πριν από την επόμενη συνάντηση των ασκιωδών ε, εισηγητών, κανονικά δηλαδή την τρίτη ε, του Στρασβούργου. 10 Μαΐου δηλαδή από τις 4 μέχρι 6 το απόγευμα. Δεν έχουν όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές προετοιμάσει τη γνωμοδότησή τους, μέχρι τότε θα πρέπει να παραλάβουμε 11 τέτοιες γνωμοδοτήσεις και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τις λάβουμε υπόψη. Οι τροπολογίες τις οποίες ε, εξετάζουμε στην παρούσα φάση είναι τροπολογίες που προέρχονται από τα μέλη της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ε, θυμίζω ότι εδώ υπάρχουν ε, ε από κοινού αρμοδιότητες σε σχέση με την έκθεση αυτή ανάμεσα σε πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές. Και έτσι όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, θα εκφραστούν και δεν θα εξαιρέσουμε τομείς όπως οι μεταφορές, ε, η πρόσβαση ε, σε υπηρεσίες υγείας κτλ. Κάποιες από τις τροπολογίες μας επικαλύπτουν θα έλεγα τις αρμοδιότητες κάποιων άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών και θα προσπαθήσουμε να τα διευκρινίσουμε αυτά στα πλαίσια των συμβιβαστικών τις οποίες θα σας καταθέσουμε. Ίσως τώρα να περάσω σε κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν κάποιο ε, ειδικό βάρος. Υπάρχουν ε, αρκετές τροπολογίες τις οποίες εγώ θα θεωρούσα, θα έλεγα σημαντικές. Καταρχάς τα δικαιώματα των παιδιών και τα δικαιώματα των οικογενειών τους, όπως επίσης και το θέμα της βίας της βάρος των παιδιών, τεκμηριωμένο από έρευνες από την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεύτερον, πολλαπλές μορφές διάκρισης, διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων είναι μορφές ε, διακρίσεων οι οποίες δεν περιλαμβάνουν κάποια μορφή ε, θα έλεγε κανείς ιεραρχία. Σαν παράδειγμα ε, τα ΙΑΜΕΑ δεν έχουν μόνο να υποστούν διακρίσεις επί τη βάση μιας συγκεκριμένης μορφής διάκρισης αλλά και για άλλους λόγους πιθανώς. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι ανάπηρες γυναίκες. Μπορεί να υφίστανται διακρίσεις για πολλούς λόγους ή οι ε, έγχρωμες λέει ομιλήτρια ε, ανάπηρες γυναίκες. Μπορεί να υφίστανται διαφορετικού τύπου διακρίσεις κάθε φορά. Πολλές φορές ε, οι διακρίσεις και τα διαφορετικά επίπεδα δεν διακρίνονται εύκολα σαν παράδειγμα το να απαγορεύει στις ε, ανάπηρες γυναίκες ε, να τεκνοποιήσουν. Αυτό είναι η λεγόμενη διασταυρούμενη μορφή διακρίσεων. Είναι μια δύσκολη έννοια, αλλά έχει σημασία να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις πολλαπλές διακρίσεις και στις διασταυρούμενες διακρίσεις. Ε, η έννοια επίσης της ε, έλογης ρύθμισης είναι κάτι το οποίο και αυτό είναι δύσκολο να κρίνει κανείς. Νομίζω ότι... I.e. denial constitutes discrimination. Ε, υπάρχουν θέματα λοιπόν σύμφωνα με και το CRPD τα οποία καλύπτουν ίσως και το θέμα της κατάλληλης μορφής ε, κατοικίας, αν θέλετε. Θα έχουμε το κείμενο λοιπόν στην Ολομέλεια του Ιουλίου έτσι ώστε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, γέρος ε, τις σκέψεις μας και της παρατηρήσεις μας. Περιμένω λοιπόν και τη δική σας συνεισφορά. Ο κύριος Κόζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κυρία εισηγητρία, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες έχουμε προχωρήσει σημαντικά ε, στο τώρα. τώρα λοιπόν υπήρχαν 183 τροπολογίες και ασφαλώς περιμένουμε και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων επιτροπών είμαι πεπισμένο ότι σε τελική ανάλυση θα καταφέρουμε στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε μια πολύ καλή έκθεση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η συνάδελφος πριν από λίγο και θα ήθελα μόνο να τονίσω κάποια περιορισμένα στοιχεία τα οποία θεωρώ, ότι είναι πολύ σημαντικά ωστόσο. Αφενός, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να προχωρήσουμε με μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά τα στοιχεία, τα δεδομένα. Υπάρχουν τροπολογίες που προτείνουν άλλα στοιχεία, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, την ενεργεία. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε αριθμητικά στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετά ε, δεδομένα από τα κράτη-μέλη και δεν υπάρχει συγκρισιμότητα ως εκ τούτου μεταξύ όλων των κρατών μέλων. Για παράδειγμα, στην τροπολογία παρελθμό 22 τίθεται ακριβώς αυτό το θέμα. Συγχωρέσαμε στην 23 τροπολογία. Ακριβώς λοιπόν αυτό είναι το θέμα στην τροπολογία παρελθμό 23. Το ζήτημα ότι τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία τα οποία ε, δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασία. Ε, ε, ανταποκρίνονται σε ένα ποσοστό, αλλά στο κείμενο το ποσοστό αυτό που αναφέρεται είναι διαφορετικό. Και αυτό λοιπόν θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και καλό μαζί με τους εισηγητές και τους σκιώδες εισηγητές να φροντίσουμε να επικαλούμαστε τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία και αυτά τα στοιχεία να χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για το πώς θέλει να αλλάξει η κατάσταση στο Ευρωπαϊκό στο Κοινοβουλίο. Επίσης θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να ελέγχουν πάντα τις ε, μεταφράσεις της γλώσσας τους. Το θέμα αυτό είναι μάλλον καινούριο για μας. Δεν είχαμε ασχοληθεί ως τώρα επισταμένος με το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν λοιπόν νέοι, όροι, ορισμοί. Για παράδειγμα, το reasonable accommodation ως έκφραση. Στην ουγγρική μετάφραση υπάρχει διαφορετική ε, έκφραση, διαφορετικός όρος για αυτό το reasonable accommodation, την κατάλληλη προσαρμογή. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό στις διάφορες μεταφράσεις οι καινούργοι όροι να μεταφράζονται σωστά. Και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους πάντα να το προσέχουν αυτό. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αφορά την χρήση των πιστοτικών ταμείων και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασκήσουμε από κοινού πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση αυτή προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρέωσεις των ΕΕ σε ό,τι αφορά τα ατμωμένα πυρία και να χρησιμοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή ε, οι σχετικοί πόροι. Και αν δεν ε, τηρούνται οι προδιαγραφές, φυσικά θα πρέπει να υποβάλλονται και κυρώσεις σε ό,τι αφορά τώρα τις διάφορες ε, τροπολογίες. Πιστεύω ότι το ΕΛΚ μπορεί να συμφωνήσει με την πλειονότητα των τροπολογιών. Φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε και ελπίζουμε να βρούμε και συμβιβασμούς με τους συναδέλφους ασφαλώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Η Μίλια Μπλίτσεβιτ Κούτε έχει τώρα το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω κι εγώ γιατί η, η έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και πιστεύω ότι με τη συνεργασία με την εισηγητρία και με τους κοιόδες εισηγητές θα μπορέσουμε να πετύχουμε καλούς ε, συμβιβασμού προκειμένου πραγματικά να συμβάλλουμε στην εφαρμογή της Σύμβασης των Εθνών για τα άτομα με αναπηρία. Θα ήθελα ε, επίσης να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες πτυχές, ε, σε κάποια στοιχεία που απασχολούν την ομάδα μας ιδιαίτερα. Καταρχάς, τα θέματα της απασχόλησης ε, είναι αυτά τα οποία μας απασχολούν όλος ιδιαίτερω και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να θέσω τη σημασία των προδιαγραφών για την προστασία της πρόσβασης στην εργασία και από, τις ε, από την διακριτική μεταχείριση. Δεν έχουν εφαρμόσει τα κράτη-μέλη πλήρως αυτή την οδηγία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αγορά εργασία και τις προσαρμογές στο χώρο εργασία. Και υπάρχουν οι ίδιοι όροι σε όλα τα κρατημέλη. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση. Γιατί αυτές είναι οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή ε, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τα άτομα με αναπηρία. Θα έπρεπε λοιπόν να καλέσουμε τα κράτη-μέλη, να τα ενθαρρύνουμε να εφαρμόσουν ε, διάφορα μέτρα προκειμένου να παροτρύνουν την εφαρμογή αυτών των ε, προδιαγραφών. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια τέτοια υποστήριξη και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ό,τι το έχουμε στο χέρι μας. Ιδάλλως, το θέμα της απασχόλησης ε, των ατόμων με αναπηρία δεν θα επιληθεί. Ένας άλλος ε, τομέας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Επιτροπή μας, είναι η κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία. Και εδώ θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ε, εστίαση, γιατί χωρίς κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία, η απασχόληση τους είναι ποσοστία πολύ χαμηλή και σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μόνοι τους και εξαρτώνται από την κοινωνική βοήθεια. Και χωρίς την κοινωνική αυτή ε, βοήθεια, πολλοί ανάπηροι θα ζούσαν κάτω από το όριο της ένδυας και δεν θα είχαν ποιοτικέ ε, κοινωνικές υπηρεσίες στη διάθεση τους. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να επισήμανθει ως έλλειψη, να αναφερθεί στην έκθεσή μας και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθυστερήσει σε ό,τι αφορά την έλεγχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την αναπηρία. Και τότε είχα καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γραπτά να προβεί στην αξιολόγηση αυτή, αλλά δεν βλέπουμε να έχει αυτό αποτελέσματα στην δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το τονίζουμε στην έκθεση. Θα πρέπει να τονίσουμε μάλλον στην έκθεσή μας καθότι θα πρέπει να μπορούμε να αξιολογούμε την κατάσταση των αναπήρων στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προβούμε στη λήψη των σωστών αποφάσεων. Άρα, συνοπτικά θέλω να τονίσω ότι στην ε, συνεργασία μας θα καταφέρουμε να προετοιμάσουμε καλές ε, συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χάρκη ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια την Helga. Stevens. Είναι ένα εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης και σας ευχαριστώ και για τις τροπολογίες σας, πολλές από τις οποίες έχουμε και εμείς συνυπογράψει. Εξετάζοντα λοιπόν τι τροπολογίε που έχουν υποβληθεί από διάφορου ευρωβουλευτέ και πολιτικέ ομάδε, πολλέ είναι θετικέ και υπάρχει κοινό έδαφο θα έλεγα 80% των τροπολογιών μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί ακούσαμε αρκετά, αλλά το θέμα των παιδιών και των γυναικών με αναπηρίες. Εμείς λέμε ότι πρέπει να έχουμε στοιχεία, συνολικά στοιχεία, κυρίως όσον αφορά την βία σε βάρος των γυναικών και κυρίως των ανάπηρων γυναικών. Επίσης θέλουμε να δούμε και την σχέση που έχει αναπηρία με τη φτώχεια και αναπηρία με την ανεργία. Γι' αυτό και έχουμε υποβάλει μια ειδική τροπολογία που έχει να κάνει με τη δικιά μου χώρα, γιατί δεν ξέρω αν το ίδιο συμβαίνει και αλλού. Στην Ελλαδία πάντως συμβαίνει και έχουμε διαμαρτυρηθεί γι' αυτό στην Επιτροπή, ότι τα άτομα με αναπηρίες, κυρίως ε, ψυχικές, δεν έχουν δικαίωμα να υποφεληθούν από την εγγύηση για την νεολαία. Κανείς δεν τους εμποδίζει μεν, αλλά το σύστημα έτσι όπως εφαρμόζεται τελικά δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε τέτοια κονδύλια. Οπότε, αν η εγγύηση αυτή προβλέπεται για όλους τους νέους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, τότε και αυτοί θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση. Δεν ξέρω όμως, επαναλαμβάνω, κατά πόσο ισχύει το ίδιο και σε άλλες χώρες μέλη όχι. Σας λέω, το σύστημα έτσι όπως εφαρμόζεται δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση. Δεν είναι απλώς ότι κάποιος τους λέει όχι, δεν σας επιτρέπουμε. Τώρα και κάποια άλλα σημεία θέλω να θίξω. Η ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρίες στη λήψη αποφάσεων και το ότι πρέπει να υπάρχει ένας διαρθρωμένος διάλογος για να εφαρμόζεται ικανοποιητικά νομοθεσία. Τώρα υπάρχει και μια τροπολογία για τη διασυνοριακή οδηγία, δεν ξέρω ποια είναι, που δεν επιτρέπει βέβαια τη διάκριση ρητά, αλλά ε, θα έπρεπε να την κοιτάξουμε περισσότερο. Και κάποια γενικά ζητήματα ότι το θέμα της αναπηρίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές και στρατηγικές μας και επίσης ότι πρέπει να ε, αναθεωρείται στοχευμένα η ευρωπαϊκή πολιτική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να μπορούμε να έχουμε και εμείς μια συνολική στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Κυρίω ε, τα παιδιά πρέπει να κοιτάξουμε με αναπηρίες σε περίπτωση που προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Στηρίζουμε πάντως την ιδέα και θέλουμε να εγκρίνουμε την οδηγία για την ίση μεταχείριση. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάω. Α, και κάτι ακόμα. Ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων με αναπηρίε. Αυτό είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται στο Στρασβούργο, για παράδειγμα, κάθε δύο χρόνια έχουμε κάτι τέτοιο, και η θέση δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Υπάρχει διάταξη της στήριξης όταν ε, μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με τον προσωπικό τους βοηθό. Ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι από αυτού εδώ. Και πάλι ευχαριστώ την εισηγήτρια και προσβλέπω σε συνεργασία μαζί της και τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαίρομαι πολύ που συζητάμε πάλι αυτό το θέμα. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί άλλωστε συμφωνώ με τα περισσότερα από όσο μας είπε η Χέλικα και την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την δουλειά και τη συνεργασία που μας προσέφερε. Προσυπέγραψα πολλές από τις τροπολογίες της. Επιτρέψτε μου όμως να τιμήσω κάποια βασικά ζητήματα που θέτω με δικές μου τροπολογίες. Το πρώτο, Θεωρώ πολύ μεγάλη σημασία την ενημέρωση για την κατάσταση των ανθρώπων με αναπηρία προς όλες τις κατευθύνσεις. Μόνο αν τα προβλήματα μας γίνουν κατανοητά, θα λάβουν καλύτερες αποφάσεις για εμάς με εμάς. Το δεύτερο, πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία μας. Η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να προσαρμοστεί και δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή που κάποιες χώρες υποφέρουν από σκληρά μέτρα που τους επιβάλλει η Τρόικα, να είναι υποχρεωμένες να κάνουν περικοπές στις κοινωνικές παροχές που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Είναι σκανδαλώδες αυτό το θέμα. Και στο τέλος, είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με τα άτομα με αναπηρία στην, στο πληθυσμό των προσφύγων το προβλέπει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν φυσιολογικά και ψυχολογικά. Φανταστείτε επιπλέον να είσαι πρόσφυγας και ανάπηρος. Πρέπει να στηριχτούν οπωσδήποτε με επιπλέον μέτρα. Σε ευχαριστώ πολύ. fertig? Dankeschön. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ε, κυρία Τατιάνα Στανόκα. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Στίβενς για την εξαίρετη δουλειά της. Είναι ένα πολύ σωροπημένο έγγραφο αυτό που μας παρουσίασε σήμερα. Τώρα και εγώ έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες προκειμένου να υπογραμμίσω κάποιες παραγράφους ακόμα περισσότερο. Πρώτα απ' όλα προτείνω να τονίσουμε τη σημασία που έχει η ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, των ίδιων των ατόμων αυτών δηλαδή, και των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν σε όλες τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της σύμβασης αυτής. Θέλω επίσης να πιστήσω την προσοχή μας και στο γεγονός ότι οι διάφορες αυτές οργανώσεις πρέπει να εκπροσωπούν διαφορετικές χώρες μέλη, γιατί τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν διαφορετική κατάσταση ανάλογα με τη χώρα στην οποία ζουν και θα πρέπει να μπορούμε να ακούμε τις ανησυχίες όλων αυτών. Θα ήθελα να έχουμε και μια χωριστή παράγραφο που να υπογραμμίζει την ανάγκη για μια εκστρατεία συνειδητοποίησης όσον αφορά την ίδια τη σύμβαση αυτή των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, προτείνουμε μια διόρθωση στην παράγραφο 6 που είναι σημαντική όταν γίνεται έκκληση στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουν μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε μορφή διάκρισης που οφείλεται σε αναπηρίες, εκεί δεν πρέπει να αναφέρουμε μόνο τις γυναίκες και τα παιδιά, αλλά και τους ηλικιωμένους με αναπηρίες. Συμφωνώ επίσης και με τις ανησυχίες της εισηγήτριας γιατί τα διευθυντικά ταμεία ε, μερικές φορές δεν χρησιμοποιούνται καλά και οδηγούν ε, σε κατάσταση δερματοποίησης. Νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν τα μέτρα τα οποία αναφέρονται από την εισηγήτρια, αλλά να διακόπτονται οι πληρωμές, να αποσύρεται η βοήθεια στην περίπτωση που διαπιστώνουμε ότι δεν γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει και όπως προβλέπονται. Τέλος για την παράγραφο 17 που ζητάει Α, όσον αφορά τα στοιχεία, τα δεδομένα που έχουμε για τους ανθρώπους με αναπηρία θα ήθελα να έχουμε ε, στοιχεία κατά περίπτωση, κατά ομάδα, δηλαδή ανάλογα με το φύλλο, την ηλικία, το αν πρόκειται για άτομα που ζουν στην Ήπεθρο ή στις πόλεις και να ξέρουμε το είδος της αναπηρίας που έχουν. Πρέπει να υπάρξει έρευνα και συλλογή δεδομένων επίσης όσον αφορά την βία και την εκμετάλλευση ανθρώπων με αναπηρίες, όποια και να είναι η αναπηρία τους. Ευχαριστούμε Λάουρα. Ατζέα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Στίβενς για την εξαιρετική της δουλειά. Και εμείς νομίζω ότι προσπαθήσαμε να συνεισφέρουμε με θετικό τρόπο έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο το οποίο να καλύπτει τους περισσότερους και να περιλαμβάνει προτάσεις αποτελεσματικές. Αναζητήσαμε να εντάξουμε όλες τις ε, τροπολογίες οι οποίες για μια στιγμή διακόπτει ο πρόεδρος για τεχνικό λόγο. Ganze, ganze Übersetzung ist weg. Hallo? Kann uns, hört uns jemand? Μας ακούτε παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος. We have no sign in the display. Is there any technician for this? Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην οθόνη. Σα <laughs> Ναι, να μιλήσουμε. Μάλιστα, πολύ ωραία που καταστάθηκε το πρόβλημα, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Τέλεια. Μάλιστα. Ακούτε λοιπόν όλοι. Πολύ ωραία. Λάουρα, έχεις το λόγο. Salto il preambolo, ringraziando la collega Steven perché ha Λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω λέει για μια ακόμη φορά η κυρία Τζέα την Στίβενς για την εξαιρετική της δουλειά. Και εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογίες. Ήρθαμε σε επαφή με τους άμεσα ενδιαφερομένους, τους ανθρώπους για τους οποίους καλούμεθα σήμερα εδώ να συζητήσουμε. Έχουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες θα ήθελα να συζητήσω με την συνάδελφο και με τους άλλους εισηγητές, ιδιαίτερα για τη γονική άδεια. Οι γονικές άδειες πρέπει να παίρνουν ειδική μορφή θα έλεγα για τους γονείς παιδιών με αναπηρία έτσι ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν τα παιδιά τους με πιο αποτελεσματικό ε, τρόπο. Ζητήσαμε επίσης την δυνατότητα διευκόλυνσης ε, πρόσβασης σε νομικές πράξεις και σε κυδαιμονίες των προσώπων με αναπηρία. Πολλές φορές στην Ιταλία η δικαιοσύνη για τα άτομα με αναπηρία καθίσταται η απονομή της ιδιαίτερος περίπλοκη. Θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε σε αυτούς οι οποίοι υφίστανται διακρίσεις στο χώρο εργασία τους να ενημερώνονται σωστά για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της δικαιοσύνης. Έχουμε ένα επίσης άλλο σημαντικό πρόβλημα τα λεγόμενα εμπόδια στον χώρο εργασίας, ζωή, σχολεία κτλ. Αυτό δημιουργεί διακρίσεις και περιθερο, περιθωριοποιεί τα παιδιά τα οποία χαρακτηρίζονται από τέτοιου είδους ε, ε, αναπηρίες. Τέτοια μηνύματα είναι απαράδεκτα από πλευρά της κοινωνίας μας. Η κοινωνία μας δεν έπρεπε να έχει τέτοιου είδους εμπόδια. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν αυτού του είδους τα εμπόδια. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με το πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά και πώς ε, θα διασφαλιστούν τα άτομα με αναπηρία στις μετακινήσεις τους. Απαιτείται λοιπόν να βοηθήσουμε, μάλλον πάλι διακόπτη, ο πρόεδρος στην ομιλήτρια για τεχνικούς πάλι λόγους. Eins, zwei, drei. kann aber gar keine Gebärdensprache. Test 1, 2, 3. are sorry, please. No, it's nothing here. Nothing on the display.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 happen. Ja, äh, Ton ist, Ton ist da, aber keine Έχουμε ήχο, αλλά δεν έχουμε σύνδεση με τις ερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Ah ja. τώρα λοιπόν έχουμε και πάλι ότι χρειάζεται. Εγώ ακούω την τερμηνία. η τερμηνείς είναι πάντα στην διάθεσή σα. Ακούτε λοιπόν όλοι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρο. Όχι πάλι από την αρχή όμω, κυρία Ετζία. Λάουρα, έχετε το λόγο onde evitare che poi si dica che io porto sfortuna. Λοιπόν, για να αποφύγουμε να πούμε ότι είμαι γρουσούζα, θα κλείσω. θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες επιλογής τις οποίες έχουν ε, τα πρόσωπα με αναπηρία γιατί τα θέματα και κάποιες έννοιες όπως αυτοί που παρέχουν φροντίδα, η φροντίδα στο σπίτι και τα λοιπά είναι θέματα στα οποία απαντήσεις ε, δεν έχουν δοθεί. Επίσης ε, κάποιες μέθοδοι εργασίας όπως το smart working και το η εξαποστάσεως εργασία δεν έχουν επίσης βρει λύσεις. Στην Ιταλία υπάρχει η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να πληρώνουν κάποια γελία πρόστιμα επειδή δεν προσλαμβάνουν αναπήρωση. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα επιπλέον πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και ένα άλλο πρόβλημα που είναι επίσης πολύ ιταλικό είναι το πρόβλημα των ψεύδοαναπήρων και ε, πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την κυρία Στίβενς. So, Πολύ ωραία. Τα καταφέραμε, λέει Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ναι, κυρία Μιλάν. Θέλω να καθησυχάσω την εισηγήτρια για το ότι θα συνεργαστούμε μαζί της όσο καλύτερα μπορούμε. Και θα σταθούμε στα θεμελιώδη ζητήματα. Εδώ, όσον αφορά την αναπηρία, υπάρχει μια παρεξήγηση. Είναι ένα γενικό όρο, ο οποίο έχει να κάνει με τόσο διαφορετικέ περιπτώσει μεταξύ του, και εξαρτάται και από τη σοβαρότητα της αναπηρίας. Πώς, ε, να το πω, από την πιο απλή αναπηρία που θα μας πλήξει όλους κάποια στιγμή στη ζωή μας. Γιατί είναι πράγματα που με την ηλικία μας συμβαίνουν. Οπότε να πούμε ότι ηλικιωμένοι οι ανάπηροι ηλικιωμένοι είναι έτσι κι αλλιώ ανάπηροι. βέβαια υπάρχουν και άλλοι που έχουν γενετικέ αναπηρίε, έτσι, γενετή. Και που για αυτού απαιτείται μια αξιοπρεπή μεταχείριση και βοήθεια. Η κοινωνία λοιπόν στο σύνολό τη, είτε πρόκειται για την ευρωπαϊκή κοινωνία είτε την εθνική, οφείλει σε κάθε άνθρωπο που έχει κάποια δυναμία στη λειτουργία του, είτε είναι ανατομικής φύσεως, είτε είναι σωματική αναπηρία, είτε ψυχο, ε, οτιδήποτε, να δίνει ό,τι βοήθεια μπορεί. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα αντιστάθμισμα με λογικά μέσα, όπως λέει και το κείμενο. Και θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε αυτό συνέχεια. Δεν πρόκειται για διόρθωση για αποκατάσταση. Αυτό είναι το πρώτο. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι όσοι βοηθούν, οι εργοδότες ή οποιοδήποτε παρεμβαίνει κάποια στιγμή για να διευκολύνει, να βοηθήσει τον ανάπηρο στη ζωή του. Είτε πρόκειται για καινοτομίε. είτε πρόκειται για start-up. Ας ελπίσουμε ότι η αναπηρία θα μπορεί από μόνη της να αποκατασταθεί, ανάλογα βέβαια με τα μέσα που διαθέτουμε, ανάλογα με τα κοινωνικά συστήματα της κάθε χώρας, αλλά και ανάλογα βέβαια με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Και φυσικά εξαρτάται από τη σοβαρότητα, έτσι από το πόσο μεγάλη είναι η αναπηρία. Το δεύτερο που συχνά συζητάμε είναι ότι η αναπηρία είναι κάτι το αντικειμενικό και ότι η διάκριση που είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε συνέχεια στη συζήτηση, είναι υποκειμενικός όρος. Αυτή τη διάκριση πρέπει να την κάνουμε και νομίζω ότι είναι ευθύνη της κάθε χώρας να φροντίσει οι ανάπηροι να μην νιώθουν θύματα διακρίσεων, εννοείται, αλλά να μπερδεύουμε τα πράγματα. και να καταλήγουμε στο γελίο, επιτρέψτε μου αυτό τον όρο, να πούμε ότι υπάρχουν πολλαπλές αναπηρίες, επειδή είμαστε φτωχοί, μετανάστες, ε, ε, γυναίκες, ε, τρανς κτλ. Νομίζω ότι εδώ βερδεύουμε τα πράγματα και το πρόβλημα το κοιτάμε από τη λάθος οπτική γωνία, γιατί δεν αντιμετωπίσουμε την πραγματική αιτία η οποία θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα ένα ευρωπαϊκό κείμενο όποια μορφή και αν έχει, να είναι αποτελεσματικό. Έτσι θα είναι αναποτελεσματικό και να μην μας εκπλήσει που οι ευρωσκεπτικιστές γίνονται όλο και περισσότεροι στην Ευρώπη. Κατά τα άλλα, κυρία Συγήτρια, να είσαστε σίγουροι ότι θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τσούρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και για τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε η κυρία Στίβεν. Ως σκιώδης εισηγητής στην Επιτροπή Μεταφορών με μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να σας μεταδώσω ότι η τεράστια πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής μου Επιτροπής έκανε δεκτή την γνωμοδότησή μας. Είναι μια εξαιρετική γνωμοδότηση, βελτιώνει νομίζω σε κάποια στοιχεία την έκθεση της Χέλγα, προσθέτει ορισμένα επιπλέον θέματα έτσι ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να μπορέσουν πλήρως να, έχουν, να βλέπουν τα δικαιώματά τους να γίνονται σεβαστά. Δίδονται ε, και κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν από τους συναδέλφους προηγουμένους. Πρέπει να υπογραμμίσουμε λοιπόν ότι υπάρχει πλήρης και πρέπει να υπάρχει πλήρης πρόσβαση ε, ενημέρωση μάλλον για την πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς όπως τα αεροσκάφη ε, και ο σιδηρόδρομος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τις εταιρείες που ασχολούνται με τις μεταφορές και αυτό περιλαμβάνει και την χρήση του αριθμού 112, 112 δεν είναι κάτι το οποίο ανακουφίζει απλά τους ε, ανθρώπους με αναπηρίες, αλλά είναι κάτι το οποίο διασφαλίζει τις συνθήκες ασφαλείας στην μεταφορά τους, στη μετακίνησή τους. Είναι μια σωστή νομίζω βάση για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο μέλλον. Ο κύριος Φουντούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με την έκθεση της συναδέλφου Στίβενς και τη συγχαίρω. Η αποδοχή των προτάσεων της έκθεσης από εμάς και των υφισταμένων νομοθεσιών της Ευρωπαϊκής ε- ε- ε- Ένωσης σχετικά με τα άτομα με αναπηρία από τα κράτη-μέλη είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον εφαρμόζονται. Δεν μπορεί στις χώρες που βιώνουν την οικονομική κρίση τα άτομα με αναπηρία να είναι ο εύκολος στόχος για εξοικονόμηση πόρων εκ μέρους των κυβερνήσεων. Στην Ελλάδα τα επιδόματα της προνοίας δεν κατάβονται. Τα οικογενειακά επιδόματα δίδονται στο 50% και τα άτομα με αναπηρία που εξαρτάται η επιβίωσή τους από αυτά τα χρήματα είναι τώρα, σήμερα σε απόγνωση. Η κυβέρνηση εχθές το βράδυ πήρε όλα τα αποθεματικά από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αφήνοντας χιλιάδες ασφαλισμένους χωρίς φάρμακα. Σας το λέγω με το λόγο της γνώσεώς μου διότι αυτό το πρόβλημα το βιώνω και εγώ ο οποίος έχω μία κόρη με ειδικέ ανάγκες και δεν υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο, από το οποίο εξαρτάται η επιβίωσή της, δεν υπάρχει στα κεντρικά φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Η Ελλάδα περνάει δύσκολες ώρες. Αυτή είναι επιλογή της κυβέρνησης και όχι υποχρέωσή της. Δεν μπορεί μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφήνει τα άτομα με αναπηρία στο έλεος της τύχης. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα αυτά έχουν δυσκολεύσει με απίστευτη γραφειοκρατία την πρόσβαση σε φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Οι γιατροί συνταγογραφούν τα απαραίτητα φάρμακα και οι υπηρεσίες μέσα από ένα δεδαλώδες γραφειοκρατικό σύστημα τους αναγκάζουν σε απίστευτη ταλαιπωρία. Η πρόσβαση στα φάρμακα, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία, έπρεπε να είναι δεδομένη. Η στήριξη των οικογενειών που έχουν παιδιά ή μέλη με αναπηρία δείχνει και τον πολιτισμό μας γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιλέξει να έχουν τα άτομα αυτά κοντά τους και να μην τα εγκαταλείπουν σε κάποιο ίδρυμα. Δυστυχώς, στην Ελλάδα της συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχουν αφαιθεί τα άτομα με αναπηρία στο έλεος του Θεού και πολλές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αρκεί να ευχαριστηθούν οι δανειστές. Σας ευχαριστώ. Danke. Μάλιστα, δεν θα κάνει άλλο το λόγο, λέει ο Πρόεδρο, και θα ήθελα λοιπόν για το λόγο αυτό να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Γκράνου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποδέχεται ιδιαίτερα ευνοϊκά την έκθεση της κυρίας Στίβενς και την ευχαριστούμε για αυτή την ε, ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συζήτηση που μπορέσαμε να έχουμε μαζί της παράλληλα με τις εργασίες αυτές. Φυσικά και στηρίζουμε το διάβημα της εισηγήτριας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε μεταφέρει τα σχόλιά μας διμερώς, αλλά εδώ θέλω να πω ότι οι πτυχές της έκθεσης που έχουν να κάνουν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μας αφορούν βέβαια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να σας πω, ότι εργάζεται πάνω σε αυτά τα ζητήματα και μάλιστα μόλις ξεκίνησε μία ενδοπηρεσίακή διαβούλευση όσον αφορά τη διαφορετικότητα και την ε, ε, αποφυγή αποκλεισμών μέσα στις υπηρεσίες. Θα δούμε λοιπόν τι θα βγει από αυτά. Οπότε αυτά δεν θέλω να σας καθυστερήσω περισσότερο. Επιβεβαιώνω λοιπόν ότι συμφωνούμε και ότι παρακολουθούμε τόσο τις συστάσεις όσο και τις επικρίσεις που περιλαμβάνει στο κείμενό της η συγγήτρια για τόσα δεν έχουν γίνει ακόμα δηλαδή είτε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είτε από τις χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι ολοκληρώσαμε και τη ζήτηση αυτή στις 30 Μαΐου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Πώς είπατε, λέει ο Πρόεδρος. Α, μάλιστα. Κύριε Στέβεντς, θέλει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο τελευταία λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες εισηγητές και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λαμβάνει γνώση και παρακολουθεί το έργο μας. Ήταν ε, θετικές οι αντιδράσεις. Πράγματι την έκθεση αυτή πρέπει να την αντιληφθούμε ως εξής. Πρόκειται για την εφαρμογή και πρόκειται και για απάντηση στις καταληκτικές παρατηρήσεις του ΟΙΕ. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε πολύ περιορισμένοι. Πρέπει να παραμείνουμε στα πλαίσια των καταληκτικών συστάσεων και τίποτα άλλο. Γι' αυτό και δεν ανέφερα όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις αναπηρίες της Επιτροπής. Απλώς είδαμε ποιες είναι οι καταληκτικές παρατηρήσεις και πάνω σε αυτές αντιδράσαμε. Γι' αυτό ίσως να σας φάνηκε μερικές φορές ότι δεν περιλαμβάνονται όλα τα θέματα όπως θα θέλατε περιλαμβάνονται, αλλά σε χωριστό κείμενο. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε τους περιορισμούς. Εδώ πρόκειται για μια έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή. Τώρα, 100% συμφωνώ με τον συνάδελφο Κόσα για τη σημασία που έχει η σωστή, η ορθή μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Η δική μου διερμηνείς ένας άκουγε την Ολλανδική καμπίνα και όταν ε, είπαμε τον όρο accommodation άκουσε στη μετάφραση housing, δηλαδή στέγαση, ενώ ε, πρόκειται για την προσαρμογή. Αυτό είναι ένα μικρό μόνο παράδειγμα του λόγου για τον οποίο πρέπει να ζητάμε από τους συναδέρφους να ελέγχουν ξανά και ξανά τις μεταφράσεις ώστε να περνάει το ορθό μήνυμα σε όλες τις γλώσσες. Βέβαια, ευχαρίστως να βοηθήσουμε κι εμείς με την σωστή ορολογία στις γλώσσες σας. Σημείωση του διερμηνέα accommodation σημαίνει και τα δύο. Για τους ηλικιωμένους τώρα, για τα παιδιά, για την νομική προστασία και για την ε, σημασία που έχει η για τις καταχρήσεις όσον αφορά τα διευθυντικά ταμεία, συμφωνώ απόλυτα. Η έννοια της αναπηρίας, θα έλεγα, είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε στα πλαίσια της υποκειμενικής έννοιας της αναπηρίας. Είναι πολύ σημαντικό να απομακρυνθούμε από την ιατρική φιλοσοφία της αναπηρίας, γιατί η αναπηρία δεν είναι μόνο η ανικανότητα να ακούει κανείς ή να περπατάει. Μπορείτε να πείτε ότι κάποιος έχει 10, 15, 70% αναπηρία. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να δείτε το περιβάλλον, τους παράγοντες, το τι συνδέει τον άνθρωπο με το περιβάλλον του και όποιος έχει περιορισμούς ή αναπηρία στο περιβάλλον που ζει αυτή η σχέση ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχει κάποια αναπηρία. Αυτή τη φιλοσοφία υποστηρίζω εγώ. Τώρα προσβλέπω στις συνεδριάσεις με τους σκιώδεις εισηγητές προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, στις 30 Μαΐου θα ψηφίσουμε εδώ στις Επιτροπή μας να ευχαριστήσω τους διερμηνείς, λέγε πρόεδρος, τους διερμηνείς της νοηματικής και ε, τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την καταγραφή ε, του κειμένου στη Γερμανία είναι κάπου και θα τα πούμε την επόμενη φορά ε, στην επόμενη συνεδρίαση στις 24 Μαΐου 2016. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και παρακαλώ τους συντονιστές να μείνουν εδώ για να ξεκινήσουμε τις με τη συνάντηση των συντονιστών. <coughs>